Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε τη μεγάλη τιμή να καλωσορίζουμε, να καλωσορίσουμε τον Ομάμ Χαμπούντι, πρόεδρο της Ιρακινής Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων. Προσεκλήθη προσωπικός από τον πρόεδρο μας, κύριο Ελμάρ Μπρόκ. Αλλά επειδή την Κυριακή διεξάγονται εκλογές στη Γερμανία, γενικές εκλογές, χρειάστηκε απρόσμενα να μεταβεί στην πατρίδα του. Και είπα ήδη στον κύριο Χαμουντή ότι θα πρέπει να αρκεστεί στην ταπεινότητά μου. Δεν υπάρχει βέβαια καμιά αμφιβολία ότι όλοι ενδιαφερόμαστε τα μάλα για τα διεξαγόμενα στο Ιράκ, τα τεκτενόμενα στο Ιράκ. Και πάνω απ' όλα μας αγγίζει η τραγωδία και η θάνατη τόσων αθών στη χώρα σας πρόσφατα. Επίσης θα θέλαμε από εσά να ακούσουμε πόσο κρίνεται τη συνέπεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία και την παρουσία ομάδων της Αλκάιντα και τζιχαδιστών στη Συρία που ενδεχομένως έχουν και κάποιες διασυνδέσεις με τη δική σας χώρα. Περιμένουμε να ακούσουμε λοιπόν τις απόψεις σας. Σας καλώ να λάβετε το λόγο για μια παρουσίαση 10-15 λεπτών και βέβαια οι συνάδελφοι στη συνέχεια θα ε, εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να ε, καταθέσουν ερωτήσεις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 πρόσκληση να συναντήσω συναδέλφους εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εν γέννη τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δράτω με τις ευκαιρίες για να απευθύνω τις ευχαριστίες μου Δράτω με τις ευκαιρίες λοιπόν για να πεθύνω τις ευχαριστήριες μου στους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γενικότερα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλους αυτούς οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό μας την ώρα που δείχναμε τα θεμέλια της δημοκρατίας και οργανώναμε εκλογές στη χώρα μας. Εγώ Παρακολούθησα όλη τη διαδικασία σύνταξης του νέου συντάγματος. Ήμουν μάρτυρας της υποστήριξης που μας προσέφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση, απτής υποστήριξης και ουσιαστικής υποστήριξης και παιδαγωγικής βεβαίως ε, προσφοράς για να βελτιώσουμε τη σύνταξη του συντάγματός μας. Το σύνταγμα του Ιράκ ήταν μια πρώτη εμπειρία θέσπισης θεμελιώδους νόμου στη χώρα μας. Μετά από αυτόν ακολούθησε η Αραβική Άνοιξη και πιστεύω ότι εμείς ήμασταν ένα παράδειγμα, ένα υπόδειγμα δημοκρατίας και ένα πρώτο βήμα στον εκδημοκρατισμό στην περιφέρεια μας. Το Ιράκ κατάφερε να εδρεωθεί ως ένα κράτος κοσμικό μου ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας του Ιράκ μπορεί να, πρόεδρος της Δημοκρατίας του Ιράκ μπορεί να εκλεγεί και, από, και μεταξύ των μη μουσουλμάνων, πράγμα το οποίο δεν ισχύει στις λοιπές αραβικές χώρες. Ε, και ως εκ τούτου εδρεώνεται και η έννοια της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπινών δικαιωμάτων, του σεβασμού του άλλου, του διαφορετικού. Έτσι λοιπόν και χάρη στις δημοκρατικές αυτές αρχές μπορέσαμε εμείς στο Ιράκ να αποτελέσουμε ένα υπόδειγμα, ένα υπόδειγμα το οποίο υπευλήθηκε προς τον Αραβικό Σύνδεσμο ε, ως ε, μοναδική, μοναδικό συνδυασμός και συγκερασμός των αρχών του Ισλάμ και της ε, δημοκρατίας. Μπορεί να αντιμετωπίσαμε σημαντικά προβλήματα. Αποτελούμε όμως ως χώρα ένα πρότυπο συνεργασίας, συνύπαρξης και μαζί με σας θα θέλαμε αυτή η εμπειρία, αυτή η συνύπαρξη να εμβαθυνθεί αλλά και να αποτελέσει πρότυπο για άλλους. Μια άλλη μοναδική εμπειρία, μοναδική για τον ε, αραβικό κόσμο, ήταν η πάταξη της τρομοκρατίας. Το Ιράκ είχε αποτελέσει ε, κέντρο συνάντησης τσιχαντιστών από ολόκληρο τον κόσμο. Από το 2006 έως το 2012 ήταν το επίκεντρο της δράσης των τσιχαντιστών και πολύ συχνά ακούγαμε από τα ε, μέσα, τα διεθνή μέσα ενημέρωση ότι θα διαμελιστεί το Ιράκ, ότι θα ξεσπάσουν πολύ εμφυλοί πόλεμοι, ότι θα μπορέσουμε να συνεπάρξουμε διαφορετικές θρησκείες και δόγματα. Τα ξεπεράσαμε όμως όλα αυτά και μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε και την τρομοκρατία. Τρίτον, η οικονομική ανάπτυξη του Ιράκ με ένα ποσοστό ανάπτυξης της τάξης του 9%, το υψηλότερο της περιφερειάς μας. Ανάπτυξη η οποία όντως στηρίζεται σε ένα μόνο σε μία μόνο πρωτοπαραγωγική πηγή το πετρέλαιο, αλλά δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι και η μεσαία τάξη ε, γνωρίζει αύξηση των εισόδων των εισοδημάτων της και ότι παρουσιάζει η οικονομία μας μια εικόνα πολύ δυναμική όπως και η κοινωνία μας γιατί βλέπουμε να γίνονται διαδηλώσεις, ε, εκδηλώσεις ε, διαμαρτυρίας, ε, δραστηριοποιούνται οι πολίτες στη χώρα μας αποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό ότι, ότι είμαστε ένας λαός με αποφασιστικότητα, αυτοπεποίθηση, ένας λαός που ξέρει τι ζητάει και θα ήθελα να μιλήσω για την ε, γεωργία. Περίπου μισό δισεκατομμύριο δολάρια δαπανά το Ιράκ σε ενισχύσεις προς τους γεωργούς του για την παραγωγή. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε αυτάρκεια σε αρκετούς τομείς της γεωργίας, δεν έχουμε καταφέρει. Αυτά για τη γεωργία. Για την εκπαίδευση, το Υπουργείο παιδείας, το, οι αρμόδιοι για τα άνωτα ιδρύματα, αφιερώνουν σε 3.000 περίπου φοιτητές ένα πολύ υψηλό ποσό για να τους υποστηρίξουν ένα ποσό περίπου 3.300 δολαρίων για έναν ε, φοιτητή μόνο του, αλλά και 3.600 για έναν παντρεμένο φοιτητή, όταν αυτό θέλει να σπουδάσει στο εξωτερικό στα εκπαιδευτικά ευρήματα. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη επίσης. Η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο Ιράκ είναι ουσιαστικά δωρεάν. Ε, για οποιαδήποτε περίπτωση δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε στα δικά μας νοσοκομεία μπορεί η κυβέρνηση να προσφέρει μέχρι 3 εκατομμύρια το μήνα, γιατί αυτό προβλέπει ο προϋπολογισμός μας, για πολίτες ασθενείς Ιρακινούς, οι οποίοι θέλουν να μεταβούν στην Τουρκία ή σε κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού για νοσηλεία. Η άντληση του πετρελαίου κυμαίνεται στο 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, παραγωγή η οποία μπορεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Παραγωγή έχουμε επίσης και σε φυσικό αέριο, αλλά αναμένουμε τις ε, άδειε, την έκδοση των συγκεκριμένων αδειών που απαιτούνται. Ένα ζήτημα που μας απασχολεί είναι η ασφάλεια, πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται τους τελευταίους τέσσερις μήνες. Ενώ είχαμε επιτύχει ένα αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας, τους τελευταίους τέσσερις μήνες έχουμε προβλήματα πάλι. Η δική μας εκτίμηση είναι ότι αυτά τα προβλήματα ασφάλειας σχετίζονται με την κατάσταση στη Συρία και κυρίως την ε, σημαντική βοήθεια που προσφέρουν ορισμένες χώρες της περιοχής μας στους εμπολέμους στην περιοχή. Ξέρετε ότι υπάρχουν ομάδες τσιχαντιστών, υπάρχουν ομάδες τρόμοκρατών του μετόπου Αλνάστρα και λοιπόν ομάδων την ε, Συρία, οι οποίοι δεν περιορίζουν τη δράση όμως μόνο στη Συρία. Την επεκτείνουν και στο Ιράκ και ως εκ τούτου ε, έχουμε συνέπειες, επηρεάζεται η κατάσταση της ασφάλειας στο Ιράκ. Ο Ισλαμικός στρατός ε, Συρίας-Ιράκ και το μέτωπο Αλνάστρα έχουν επηρεάσει σημαντικά την κατάσταση στο Ιράκ. Έχουν μεγάλη απήχηση, έχουν την υποστήριξη του Κατάρ αρχικά, στη συνέχεια της Σαουδικής Αραβίας, η οποία ανέλαβε τη σκητάλη, κυρίως ε, στο πρόσωπο του πρίγκιπα Μπαντάρ έχουν βρει υποστήριξη. Και ως εκ τούτου εμείς αντιμετωπίζουμε σημαντικά προβλήματα ασφάλειας. Παραδείγματι η επίθεση στη φυλακή Ρούμπερ με συνέπεια την απελευθέρωση 500 ε, τρομοκρατών και σημαντικές επιθέσεις ε, που γνωρίζουν γεωματρική άνοδο τον τελευταίο καιρό. Θα έχετε ενημερωθεί ασφαλώς ότι καθημερινά έχουμε έκρηξεις βομβών με δεκάδες θύματα η επιμελητία που έχουμε στη θέσή μας δεν, είναι απεριό, δεν έχει απεριόρους τους σπόρους ε, και ε, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε παγιδευμένα αυτοκίνητα σε δημόσιο χώρο και με, τηλεκατευθυνόμενη, με τηλεκατευθυνόμενο μηχανισμό δεν είμαστε θέση να τα αντιμετωπίσουμε. Έχουμε πολλές φορές ε, επιθέσεις αυτοκτονίας σε κηδείες ή άλλες εκδηλώσεις μαζικές που οργανώνονται στη χώρα. Αυτές οι τρομοκρατικές επιθέσεις δεν έχουν ε, ε, σημειώσει θύματα μεταξύ αλλοδαπών ή δεν έχουν δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία ξένων επιχειρήσεων ούτε και στην ε, οικονομία της χώρας. Μέσω όμως αυτών των επιθέσεων βλέπουμε να γεννιέται ένα νέο δεδομένο στην πολιτική κατάσταση στη χώρα Και αυτό είναι οι ε, σχέσεις, η συνεννόηση, η επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων τμήματων της κοινωνίας μας και το πόσο μπορούν αυτά να επηρεαστούν από την τρομοκρατία. Από την αρχή δηλαδή της, της, ε, του σχηματισμού κυβέρνησης, από το 2010 λίγο πολύ, και από την εποχή που οι φίλοι της λεγόμενης Ιρακινής λίστας, οι Σουνίτες φίλοι μας, που ε, εκπροσωπούνται κυρίως στη δυτική χώρα, ανέλαβαν υπουργεία, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο ε, Ηλεκτρικής Ενέργειας, το Υπουργείο Γεωργίας, Βιομηχανίας, Υπουργείο ε, Οικονομικών Εθνικής Οικονομίας, το Υπουργείο Αμήνης. Μία συμμαχία λοιπόν για όλη τη χώρα, για ολόκληρο το έθνος και ασφαλώς θα αναγνωρίσετε ότι πρόκειται για Υπουργεία Κλειδιά, πολύ σημαντικά Υπουργεία, μεγάλη σημασίας, ιδιαίτερα για την εξέλιξη στη χώρα, της στη χώρα. Το Υπουργείο λοιπόν Εσωτερικών, το Υπουργείο Αμήνης παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα διότι δεν έχει αναλάβει καθήκοντα ο ε, Υπουργό δεν έχει ρυθμιστεί δηλαδή η ανάληψη καθηκόντων και έτσι έχουμε ακόμα συνεχιζόμενες εντάσεις και τριβές. Ο κύριος Χασιμή έχει εμπλακεί, κυρίως όσον αφορά το Υπουργείο των, ε, της Εθνικής Οικονομίας και τι μήνυμα αντλούμε από όλα αυτά. Το μήνυμα το οποίο αντλείται είναι ότι οι Σουνίτες φίλοι έπεσαν θύματα χειραγώγησης από ορισμένου σουλεμάδες, από ορισμένου δηλαδή ε, θρησκευτικούς ηγέτες ε, από την περιοχή Σαλαχαντίν, αλλά και άλλες περιφέρειες της χώρας. Και έτσι οργανώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις, διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, τις οποίες δεν μπόρεσε αμέσως να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, η οποία όμως στη συνέχεια ε, θέσπισε μία Διυπουργική Επιτροπή υπό τον Σάιμπουτ Λουκ, δόκτωρα Σάιμπουτ Λουκ, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Και βέβαια εκεί συζητήθηκε και το θέμα της, ε, των, των φυλακών και της ε, ισορροπίας δυνάμεων και της ε, κατάστασης σχετικά με τον ΠΑΘ. Δημιουργήθηκε μάλιστα, συστήθηκε μάλιστα μέσα στο Κοινοβούλιο μια ειδική επιτροπή για την ε, μελέτη και εξέταση αυτής της κατάστασης και των ισορροπιών στη χώρα. Όταν λοιπόν υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα, ε, είναι το έδαφος γόνιμο για την ανάπτυξη επιθέσεων τρομοκρατικών. Η πρώτη περιφέρεια στην οποία εκδηλώθηκαν αυτές ήταν η περιφέρεια Ρουμαντή, σουνετική περιοχή, από την οποία είχε εκδιωχθεί η Αλκάιντα. Αλλά και θα ήθελα να σημειώσω εδώ ότι σε σχέση και με το Ιράκ και με την ε, Συρία δεν ε, σημειώνονται αντιστάσεις επαρκής από πλευράς των ε, κατοίκων στις περιοχές αυτές κατά των τρομοκρατικών αυτών οργανώσεων ε, και ομάδων. Στο παρελθόν έδειχνε μεγάλη αντίσταση ο λαός μας στην τρομοκρατία, αλλά τώρα φαίνεται να μην αντιστέκεται και να κυκλοφορούν ελεύθερα στις περιοχές αυτές, ιδιαίτερα όπως είπα λόγω της κρίσης στη Συρία, η οποία έχει καθοριστικό ρόλο στην, κρίση, στην κατάσταση στο Ιράκ. Βεβαίως παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στη Συρία σε όλο το μήκος των συνόρων μας. Παρακολουθούμε ποια είναι η κατάσταση και οι κινήσεις των ε, φατριών και προσπαθούμε να ε, αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν πιο επιτυχώς την κατάσταση. Εμείς φυσικά τασόμαστε με το πλευρό του ε, λαού της Συρίας, να έχει την ελευθερία να επιλέξει τον ηγέτη του, ε, και ένα δεύτερο σημείο για τη Συρία θα ήθελα να επισημάνω ότι τα σώμεθα ανεπιφύλακτα κατά της χρήσης βίας. Είτε αυτή πρόκειται από το, οι καθεστωτικές δυνάμεις είτε από την αντιπολίτευση. Επίσης, τα σώμεθα ανεπιφύλακτα κατά του εμπάργου και του αποκλεισμού, του οικονομικού αποκλεισμού. Επίσης, τα σώμεθα ανεπιφύλακτα κατά της ω χημικών όπλων και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ε, δραστηριοποιηθούν τα διεθνή μέσα, τα μέσα της διεθνούς κοινότητας. Τέταρτον, ε, τα είναι επιφυλάκτα κατά των ε, αεροπορικών πληγμάτων γιατί μπορεί κανείς να δει πότε μπορεί να ξεκινήσει ο πόλεμος αλλά δεν μπορεί ποτέ να προβλέψει πότε και πώς θα τελειώσει και πιστεύουμε ότι θα πρέπει ο διάλογος να περάσει από μια μεταβατική φάση με τον διορισμό μιας μεταβατικής κυβερνήσεως η οποία θα οργανώσει εκλογές για τον, την ανάληψη καθηκόντος μιας νέας κυβερνήσεω στη συνέχεια δημοκρατική. και βέβαια ένα φύλλο πορεία για τη Συρία αλλά και ολόκληρη την περιοχή που θα ε, θέσει επιτέλους ένα τέρμα στην ε, ε, επιδίνωση το, της καταστάσεως την οποία αντιμετωπίζουμε. Οι ομάδες αυτές, οι τζεχαντιστές, οι τακφυριστές που υπάρχουν, δραστηριοποιούνται στη Συρία και οι οποίοι την χάνουν οικονομικής υποστήριξης από κάποιες άλλες δυνάμεις, θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι κινδυνεύουν, ότι ε, θέτουν μάλλον σε κίνδυνο ολόκληρη την κατάσταση και ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Όπως ακριβώς είχε συμβεί με το Αφγανιστάν. Έχουμε κάνει τις προσπάθειές μας λοιπόν, ήδη έχουμε δει μια θετική ανταπόκριση από την ε, Τουρκία, θα αναλάβουμε διαβήματα και σε σχέση με τις χώρες του Περσικού και Πιστεύουμε ότι θα πρέπει ε, να ε, δραστηριοποιηθεί η διπλωματία, η κοινοβουλευτική οδός, η ανταλλαγή επιστολών και η επικοινωνία για την επίλυση των προβλημάτων. Υποστηρίζουμε τον κύριο Μπραχήμη και την πρωτοβουλία της Γενέβης 2 σε όλες τις προσπάθειες. Είμαστε υπέρ της πρόσφατης συμφωνίας για την ε, ξέβρεση μιας ρύθμισης για τη Συρία με διαφύλαξη και αποδοχή των διεκδικήσεων του λαού της Συρίας και με στόχο την ειρήνη στην περιοχή. Αυτές είναι οι σκέψεις μας σε σχέση με το Ιράκ, σε σχέση με την ευρύτερη περιφέρεια και την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στη χώρα μας. Και βέβαια είμαι στη για κάθε ερώτηση. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Χαμουντή. Θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους ε, για το εξή. Στι 5 παρατέταρτο θα έρθει ο Πρωθυπουργό τη Αλβανία που έχει πάρα πολύ σφιχτό πρόγραμμα και ο ίδιο και ανηλυμένε υποχρεώσει. Παρακαλώ, 1,5 λεπτό έκαστο για την ερώτησή σα. Πρώτο ο κύριο Σαλαφράγκα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, καλωσορίσατε στην Επιτροπή Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολλά μέλη της Επιτροπής μας Έχουμε δηλώσει το ενδιαφέρον να, να συναντηθούμε μαζί σας και να συζητήσουμε με τους συναδέλφους μας από το Ιράκ για τις σχέσεις μας στις αμοιβές. Υπό την έννοια αυτή σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις εξηγήσεις που μας δώσατε και την περιγραφή της κατάστασης στη χώρα και νομίζω θα ήταν επιθυμητό να μπορούμε λίγο να εμβαθύνουμε σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική κατάσταση και τη συνεργασία αυτή τη στιγμή την κυβερνητική μεταξύ Σιητών και Σουνιτών να δούμε σε ποιο βαθμό το γεγονός ότι δεν έχουν διωθεί αυτά τα χαρτοφυλάκια, τα τόσο σημαντικά που είναι της άμυνας και των εσωτερικών, μπορεί να βοηθήσει να αντιμετωπιστεί η τόσο σοβαρή κατάσταση και το πρόβλημα της βίας. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, είδαμε το 2013 ήταν πάνω από 50.000 οι δολοφονικές απόπειρες, πάνω από 20.000 οι ε, τραυματίες και ε, τον Αύγουστο ήταν πολύ νεκρός ο με πάνω από 800 νεκρούς και άλλα θύματα. Ε, λοιπόν, θα μας ενδιέφερε να δούμε λίγο αυτή την ανάλυση και πώς είναι η σχέση σας ε, με τους Κούρδους στη χώρα σας και σε ποιο βαθμό επηρεάζουν και οι Σύριοι πρόσφυγες Ακούσαμε ότι είστε αντίθετοι με τη σύγκρουση, αλλά έχετε υποδεχτεί πάνω από 250.000 Σύρους πρόσφυγες. Και ε, μπορείτε να μας πείτε ε, για τα ε, εκτρά αυτά που συνέβησαν στο κάμπ Ασράφ, στο στρατόπεδο που πέθαναν πάνω από 50 και, που, και άλλοι υφίστανται ακόμα δεινά και κρατούνται. Η κυρία Κρόμπερ που είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας με το Ιράν παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλωσορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ ξέρετε είμαι πρόεδρος της αντιπροσωπείας για το Ιράν και προσπαθήσαμε να καλλιεργήσουμε και τις διακοινοβουλευτικές σχέσεις μας με το Ιράν. Ε, ποιες είναι οι δικές σας σχέσεις και η στρατηγική εταιρική σχέση που έχετε με το Ιράν. Αν θέλετε να αναφερθείτε σας παρακαλώ και να μας παρουσιάσετε και την ε, μελλοντική προοπτική. Στο Ιράν έχει εκλεγεί τώρα ένας νέος πρόεδρος και θα ήθελα να ακούσω την αξιολόγησή σας ε, για το πώς αλλάζει τις πολιτικές στη χώρα και αν υπάρχει κανένα παράθυρο ευκαιρίας, όπως λέγεται, να συνεργαστείτε, να επιλύσετε ενδεχομένω και το πυρηνικό ζήτημα. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Chairman, over here. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάνοκ, εδώ είμαι. Ε, τρεις ερωτήσεις σύντομα. Πρώτη, Ποιες δράσεις θα αναλάβει η κυβέρνηση του κυρίου Μαλίκη μετά τη σφαγή στο κάμπα 52 κρατουμένων και ε, όπου ενέχονται δεχομένω και οι ε, δυνάμεις ασφαλείας. Ε, δεν ξέρω, ρωτώ, γιατί βλέπουμε ε, και δημοσιεύματα και ανακοινωθένα από το Κοινοβούλιο. Για τη Συρία και την υποστήριξη της κυβέρνησής σας στον Ασάτ, ε, ε, στα πλαίσια του Αραβικού Συνδέσμου, σήμερα πώς βλέπετε τη δεύτερη διάσκεψη στη Γενέβη και τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτικών και Ρωσίας για ε, την καταστροφή των όπλων μαζικής καταστροφής που ε, ε, έχει πλέον αποδεχτεί και ομολογήσει ότι διαθέτει η κυβέρνηση Άσαντ που μέχρι πριν από λίγες μέρες το διέψευδε αλλά τώρα το παραδέχτηκαν. Ο κύριος Άσαντ λοιπόν θα συμμορφωθεί και θα ανοίξει το δρόμο ε, για μια ειρηνική επίλυση αυτού του ιδεχθούς εμφυλίου πολέμου. Και σε σχέση με αυτό που ρώτησε ο συνάδελφος Σαλαφράνκα σχετικά με το Κουρδιστάν. Ε, πώς αντιδρά ε, η κυβέρνησή σας ε, με την de facto περίπου ανεξαρτητοποίηση της περιοχής της κυβέρνησης του Ερμπίλ υπό την ηγεσία του κυρίου Μπαρζανή υπάρχει κανένας κίνδυνος διαμελισμού του Ιράκ έτσι, ως ενιαίο κράτος θα ήθελα να σας πω ότι πιέζει ο χρόνος και έχουμε κλείσει τον κατάλογο θα παρακαλέσω τώρα τον κύριο Βούλιανιτς Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ είμαι Κροάτης, ξέρετε, ε, που ήταν τμήμα της πρώην Ιουκοσλαβίας. Και είχαμε πολλούς φοιτητές από το Ιράκ τότε. Η χώρα εξελίσσεται από ό,τι φαίνεται τώρα και οικονομικά και κοινωνικά. Δεν υπάρχουν δεν υπήρχαν ε, συγκρούσεις ε, θρησκευτικέ. Όλα αυτά συνέβαιναν τότε. Δεν ξέρω τι έγιναν οι περισσότεροι πρώην φοιτητές μου. Ελπίζω να ζουν οι άνθρωποι και να είναι καλά. Ε, εν πάση περιπτώσει, το Ιράκ πιστεύω ότι έχει πολλούς νέους καλά μορφωμένους που μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα και να την οθήσουν σωστή κατεύθυνση. Γιατί τι τους εμποδίζει λοιπόν οι προτεραιότητες ποιες είναι για τα ζητήματα που εκκρεμούν πριν δοθεί αυτή η όθηση από τον αξιόλογο αυτό πληθυσμό νέων. Η παρουσία της Αλκάιντα αυτή, τα κατάλοιπα, τα σταγονίδια του παλιού καθεστώτος, η αντίσταση στους Αμερικανούς ή τίποτα άλλο. Ή μήπως έχει γίνει ήδη αυτή η όθηση και δεν την έχουμε αντιληφθεί. Ευχαριστώ. Ο κύριος παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ε, με ενεθάρρυναν τα όσα σαφή είπατε κατά των εξορμιστικών ομάδων και ε, σχετικά με την πολιτική της κυβέρνησής σας για να διευκολύνετε τους φοιτητές να σπουδάζουν στο εξωτερικό. Πρώτον, θέλω να ρωτήσω κάτι για την εθνική ενότητα. Υπήρξε η συμφωνία του Ερμπίλ για την ε, συνεργασία πριν από λίγα χρόνια. Τι ακολούθησε, εφαρμόζεται αυτή Εγκρίθηκε νόμος για το πετρέλαιο. Τι γίνεται με τις άλλες μειονότητες, με τους χριστιανούς. Γιατί οι περισσότεροι έχουν ε, αποχωρήσει από τη χώρα. Επίσης, στον τύπο βλέπουμε πολλά δημοσιεύματα που ισχυρίζονται ότι Ιρανικά αεροπλάνα πέρασαν από τον εναέριο χώρο του Ιράκ για να ε, δώσουν όπλα στη Συρία. Ισχύει αυτό. Παρακαλώ, κυρία Ντεμαρτίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δέκα χρόνια μετά την στρατιωτική επέμβαση που απελευθέρωσε τη χώρα από τη δικτατορία του Σαντάμ Χουσεϊν, το Ιράκ έχει επιτελέσει πρόοδο, αλλά δυστυχώς γίνονται πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις για θρησκευτικούς λόγους. Ε, η κατάσταση στη Συρία επιτείνει αυτό το εσωτερικό πρόβλημα, διότι ξέρουμε ότι πολλοί χριστιανοί ε, αποχώρησαν από τη Συρία. Εκεί διατρέχουν κίνδυνο και πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε για να επιλύσετε τις εσωτερικές ε, διαμάχες που υπάρχουν μεταξύ Σουνιτών, Σιητών και Κούρδων. Πέτερλε, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, επιμείνατε στις προσπάθειες προσπάθειες που γίνονται για την εθνική συμφιλίωση σε επίπεδο κυβέρνησης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις για τον διαπολιτισμικό και ε, διαθρησκευτικό διάλογο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χαμούντι, έχετε 15 λεπτά στη διάθεσή σας για να μας απαντήσετε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους βουλευτές που υπέβαλαν ερωτήσεις. αλλά δεν υποβάλλατε ερωτήσεις για τη σχέση μεταξύ Ιράκ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σχέση οικονομικής εταιρικής συνεργασίας μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μία συμφωνία η οποία ε, βοηθά και τα δύο μέρη. Γι' αυτό θα πρέπει να περάσουμε στην εκτέλεση αυτής της συμφωνίας. Θα πρέπει λοιπόν οι σχέσεις μας να σταθούν παραδειγματικές. Πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μία αναδυόμενη δημοκρατία που είναι το Ιράκ. Θα πρέπει να δώσουμε νέα όθηση σε αυτή τη συμφωνία. Υποβάλλατε ερωτήσεις επί της ουσίας. Και γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται. Γιατί ζούμε σε ένα παγκόσμιο χωριό κατά κάποιο τρόπο. Όσον αφορά το πρόβλημα της διένεξης μεταξύ Σουνιτών και Σιητών, θα ήθελα να σας πω ότι η κατάσταση δεν είναι ίδια αν τη συγκρίνουμε με το Ιράν, ε, Λίβανο, Αφγανιστάν ή Πακιστάν. Δεν πρόκειται για, για την ίδια διένεξη. Οι Σουνίτες και οι Σιήτες του Ιράκ ανήκουν στην ίδια φυλή. Άρα η κρίση που άρχισε μετά από την απόσυρση του ραφε Αλ Ισάουι, του Υπουργού, του Υπουργού Οικονομικών, δεν αποτελεί την πηγή της ε, ε, διένεξης. Αποφάσισε να αποχωρήσει. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι ε, ο επικεφαλής αυτής της φυλής της ε, φυλής του Υπουργού, ο οποίος ε, υπέβαλε την παρέτησή του. Ο, επικεφ... ο επικεφαλής είναι ΣΥΙΤΙΣ και ζει στην πόλη Σεντανάζεφ. Ζει στην ιερή πόλη Νάζαφ. Άρα πρόκειται για την ίδια εθνότητα για την ίδια φυλή. Όλοι ανήκουμε στην ίδια φυλή, μερικοί είναι Σιήτες, άλλοι Σουνίτες. Στη φυλή Σούμαρ ή ε, Σίναρ Ζουμπούρ πρόκειται για φυλές ε, όπου συμμετέχουν και Σουνίτες και Σιήτες και γίνονται και γάμοι μεταξύ των μελών αυτής της φυλής, έτσι ώστε να επιτυκνύουμε και κοινωνική αλληλεγγύη όταν χρειάζεται, όταν κάποιος αρρωστήσει, τότε όλοι συνεισφέρουν χρηματικά για να βοηθήσουμε το τον εν άνθρωπο. Το πρόβλημα λοιπόν μεταξύ Σιτών και Σουνιτών δεν είναι ένα πρόβλημα ε, διένεξης εθνοτήτων. Εμείς ε, δίνουμε μαθήματα στην Συρία, στο Μπαχρέν και στη Σαουδική Αραβία για να ξέρετε τι μπορεί να κάνει το Ιράκ για την συνύπαρξη των ε, διαφόρων θρησκειών. Γνωρίζετε τον Ιμάμ Αλσιστάνη, τον ε, Αγιατολάχ Αλσιστάνη. Πρόκειται για την ανώτατη αρχή για τους ΣΥΙΤΕΣ. Είπε ακριβώς ότι θα πρέπει να λέμε, να μην μιλάμε μόνο για τους αδελφούς ε, Σουνίτες, εσείς να μιλάτε για τους ε, Σουνίτες σαν να επρόκειτο για εσάς τους ίδιους. Εμείς έχουμε ένα θέμα διαχείρισης, όχι θρησκευτικής ε, διένεξης. Υπήρχε παλαιότερα συγκεντρωτισμός, ένα κόμμα ε, ένας δικτάτορας. Τώρα όμως είμαστε μια αποκεντρωμένη χώρα. Γι' αυτό υπάρχουν ε, προβλήματα στον τομέα καθαρά της διαχείρισης. Υπήρξε υπουργική κρίση η οποία όμως θα επιληθεί. Τον επόμενο Απρίλιο θα διενεργηθούν εκλογές και νομίζω ότι αυτές οι εκλογές θα μας επιτρέψουν θα επιτρέψουν να επαναπροσδιορίσουμε τον πολιτικό χώρο. Δεν υπάρχει πρόβλημα διένεξη μεταξύ Σουνιτών και Σιητών. Ο ε, Αλασάντ προώθησε τα συμφέροντα των Σουνιτών. Ε, μετέβη στο Ερμπίλ για να προωθήσει τα συμφέροντα των Σουνιτών. Στο Νότατο Συμβούλιο συμμετέχουν και οι ΣΥΙΤΕΣ. Γι' αυτό σας λέω ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι καθαρά διαχειριστικό. Υπάρχουν περιφέρειες οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, αλλά μην νομίζετε το πρόβλημα του Ιράκ αφορά ε, ένα θέμα διένεξης μεταξύ Σιτών και Σουνιτών. Βεβαίως υπάρχουν ορισμένες μορφές διάκρισης σε ορισμένες περιφέρειες οι διοικητικά διαμερίσματα, αλλά δεν αφορά τους Σουνίτες αποκλειστικά, μπορεί να αφορά και τους Σιήτες. Υπάρχει μια περιφέρεια Σιητών στο Νότο που βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Το πρόβλημά μας είναι ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση και ανησυχούμε για την ε, διοίκηση της χώρας. Τώρα θα ήθελα να σας μιλήσω για τους Σύριους πρόσφυγες. Υπάρχουν κονδύλια, 10 εκατομμύρια δολάρια έχουν ε, διατεθεί σε αυτή την ε, περιοχή του Κουρδιστάν για να μπορέσουμε να υποδεχτούμε τους πρόσφυγες. Όσο αφορά τον καταβλισμό Ασράφ, ξέρετε ότι ζητήθηκε από τους κατοίκους του Ασράφ να αποχωρήσουν από αυτό τον καταβλισμό για να μεταβούν σε μια περιοχή η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στο αεροδρόμιο. Το Ασράφ βρίσκεται σε μια περιφέρεια όπου υπάρχουν και Σιήτες και Σουνίτες, αλλά δυστυχώς και θερμοκράτες. Η Διάλα αποτελεί ένα ε, θερμό σημείο. Η Διάλα είναι μια περιφέρεια όπου υπάρχουν πολλοί κλειδονισμοί. Γι' αυτό η κυβέρνηση ζήτησε από τους κατοίκους του Ασράφ να αποχωρήσουν από τον καταβλισμό, διότι δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλειά τους. Υπάρχουν και άλλες ε, θερμές περιοχές ε, του Ιράκ, δηλαδή η περιοχή του Αμπουγκράιμπ, την οποία δεν ελέγχουμε. Δεν μπορούμε να, να υπερασπιστούμε τους κατοίκους του Αστράφη. Γι' αυτό ζητήσαμε να μεταβούν σε έναν άλλο καταβλισμό κοντά στη Βαγδάτη, υπό αμερικανική διοίκηση. Πρόκειται για κατοίκους που δεν θέλουμε να κρατήσουμε εκεί διότι ήταν και πρώην συνεργάτες του καθεστώτος του Σαντάμ Χουσέιν που είχαν σκοτώσει και Σουνίτες και Σιήτες και Κούρδους. Και πολλές φορές η αστυνομία απαγορεύει πρόσβαση σε αυτές τις γειτονιές. Εάν ένα αυτοκίνητο μπει σε αυτή τη θερμή περιοχή Ποιος ε, θα είναι ο υπεύθυνος, ε, οι κάτοικοι ή η αστυνομία που έδωσε την άδεια διέλευσης σε αυτή την επικίνδυνη περιοχή. Αυτό είναι και το ουσιώδες πρόβλημα. Η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει θέματα ασφαλείας σε καθημερινή βάση. Αντιμετωπίζουμε, έχουμε νεκρούς σε καθημερινή βάση. Οπωσδήποτε εκφράζουμε την ανησυχία μας και τη λύπη μας για όσους μεταβαίνουν στον καταβλισμό Ασράφ. Αλλά η κυβέρνηση δεν μπορεί να εξασφαλίσει την προστασία των κατοίκων στον καταβλισμό Ασράφ. Το ίδιο ισχύει και με τις φυλακές του Αμπουγκράιμπ. Ήρθαμε σε επαφή με τα Ηνωμένα Έθνη έτσι ώστε οι εκπρόσωποι τους στη Βαγδάτη να μπορέσουν να διενεργήσουν μια έρευνα για να δούμε κατά πόσο στη διαδικασία νεκροψίας μπορούμε να ε, διαλευκάνουμε υποθέσεις. Υπάρχουν χώρες όπως ο Καναδάς και η Αυστραλία που ζήτησαν να υποδεχτούν αυτούς τους κατοίκους του καταβλισμού Αστραφ. Γιατί δεν το κάνουν έμπρακτα όμως γιατί, δεν, γιατί πρέπει εμείς να αναλάβουμε αποκλειστικά την ευθύνη. Νομίζω χώρες όπως η Αυστραλία και ο Καναδάς θα μπορούσαν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Στο Ιράκ υπάρχουν διάφορες εθνότητες και θρησκεύματα, Κούρδοι, Σιήτες και Σουνίτες. Αυτό αποτελεί και μία πηγή ευκαιριών θα μπορούσαμε όλοι να υπηρετήσουμε το ε, Ιράκ και την ευρύτερη περιφέρεια. Εμείς δεν υποστηρίζουμε το Ιράν και δεν μπορούμε να υπηρετούμε τη Σαουδική Αραβία διότι το άλλο ημισή του πληθυσμού δεν θα συμφωνούσε. Δεν μπορούμε να υπηρετούμε τη ΣΥΠΑ διότι το ημισή του πληθυσμού δεν θα το υποστηρίζει. Εμείς θέλουμε να έχουμε σχέσεις με όλο τον κόσμο και υπάρχει μία ε, μειονότητα από το Τουρκμενιστάν που θα μπορούσε να αποτελέσει γεφυροποιό στοιχείο με την Τουρκία. Το ίδιο αφορά και την ε, Σαουδική Αραβία. Μπορεί να υπάρξει μία διαδικασία γεφύρωσης ή προσέγγισης. Μπορούμε να έχουμε λοιπόν σχέσεις με ολόκληρο τον κόσμο. Υπάρχουν και σχέσεις ε, Ιράκ και ΙΠΑ. Εμείς θα μπορούσαμε να διαμεσολαβήσουμε στην περίπτωση του Ιράν. Μπορούμε να διαβάσουμε μηνύματα. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου μας επισκέφτηκε την Τουρκία και στο εγγύς μέλλον θα μεταβεί στη Σαουδική Αραβία έτσι ώστε να αποκατασταθούν οι σχέσεις, να οικοδομηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης. Η της Βαγδάτης θα είναι το αντίστοιχο της Γενέβης σε θρησκευτικά ζητήματα. Δηλαδή οι πολιτικοί άνδρες, οι προσωπικότητες αυτές θα μπορέσουν να προσφέρουν τις καλές ναι. τους υπηρεσίες και υπάρχουν ε, σχέσεις ε, προς όλες τις κατευθύνσεις. Έτσι εμείς βιώνουμε και βλέπουμε το νέο Ιράκ που θα μπορούσε να είναι ένας παράγον σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και ε, μία γέφυρα μεταξύ όλων των ε, εμπλεκομένων μερών. Να γεφυρώσει τις ε, διαφορές ως προς τον νέο πρόεδρο του Ιράν γνωρίζουμε ότι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο ως προς σχέσεις με τη Δύση και θα μπορέσει να συνεισφέρει να επιλύσει και το θέμα των πυρηνικών, καθώς και άλλα. Δεν υποστηρίζουμε τον Αλασάντ, είμαστε υπέρ της μετάβασης σε ένα δημοκρατικό καθεστώς στη Συρία. Τα αεροπλάνα που χρησιμοποίησαν τον εναέριο χώρο μας ε, υπέστησαν ελέγχους. Ερευνήθηκαν και έχουμε έρθει σε επαφή και με την αντιπολίτευση της Συρίας. Συμφωνούμε με τη Γενέβη 2, υποστηρίζουν τις καλές υπηρεσίες του κυρίου Λάκτα Ιμπραχήμ, ε, καταδικάζουμε τη χρήση χημικών όπλων διότι ήμασταν και το πρώτο θύμα χρήσης χημικών στο Ιράκ όπως γνωρίζετε. Και Θα ήταν πολύ χρήσιμο ε, να μην είχε γίνει, να είχαμε χρησιμοποιήσει τις καλές υπηρεσίες των ε, διαμεσολαβούντων όταν εμείς ε, υποστήκαμε την χρήση, την, τα, χημικά όπλα, τη χρήση αυτή των χημικών όπλων, όταν εμείς υπήρξαμε τα πρώτα θύματα χρήσης των χημικών όπλων. Δεν νομίζω ότι το Κουρδιστάν επιθυμεί τον διαχωρισμό του. Τον διαχωρισμό από το έδαφος μας. Πιστεύω ότι οι διάφορες περιφέρειες χρησιμοποιούν δίκαια τα έσοδα από το πετρέλαιο και αυτό αποτελεί ενωτικό στοιχείο όπως και το φιλετικό στοιχείο, όπως σας είπα στην αρχή της εισήγησής μου. Δεν νομίζω ότι ε, υπάρχει μέλλον για αυτή την αυτονόμηση και δεν θα ήταν και ευκταίο. Σε σχέση με τους φοιτητές στην Κροατία ή τη Ρουσία θα ήθελα να πω ότι και οι φοιτητές διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο μεσολάβησης. Το Ιράκ βρίσκεται σε καλό δρόμο, υπάρχουν βεβαίως προσκόμματα και επιφυλάξεις κατά του αναδιόμενου αυτού δημοκρατικού καθεστώτος, αλλά προχωρούμε με μικρά βήματα και βεβαίως ε, ανησυχούμε ιδιαίτερα για τις χώρες του κόλπου και για την κατάσταση στη Συρία. Με τη βοήθεια του ε, Θεού θα τα καταφέρουμε. Όσον αφορά την ε, μειονότητα των χριστιανών, θα ήθελα να σας πω ότι βάσει του συντάγματός μας όλες οι μειονότητες την χάνουν προστασίας. Ε, χαίρουν όλων των δικαιωμάτων και αυτό αφορά και τους χριστιανούς. Ε, ζουν το χρυσό αιώνα, ζουν ένα χρυσό αιώνα αυτές οι μειονότητες, εξαιτίας μάλλον χάρη του νέου συντάγματος. Δηλαδή οι Ιρακινοί μπορούν να κατακτήσουν όλα τα ε, αξιώματα κάτι το οποίο δεν ισχύει σε άλλες μουσουλμανικές χώρες. Δηλαδή το Σύνταγμα επιτρέπει σε έναν χριστιανό να κατέχει ακόμα και τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν υφίστανται καμία διάκριση οι χριστιανοί, ούτε οι Κούρδοι. Δηλαδή οι χριστιανοί ε, δυστυχώς πλήττονται από αυτά τα, ε, αυτές τις τρομοκρατικές δράσεις, αλλά εξίσου όπως όλοι οι άλλοι, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Οι Σιήτες έχουν ε, υπάρξει τα σοβαρότερα θύματα αυτής της ε, τρομοκρατικής ε, δράσης. Και αυτό το βλέπουμε με βάση τα αριθμητικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να μας βοηθήσει σε αυτή μας την ε, πορεία και να προτείνει και επιμορφωτικά προγράμματα για τους υπαλλήλους μας. 3.000 ε, υπάλληλοι έχουν ε, μεταβεί στην Ιαπωνία για κατάρτιση, επιμόρφωση και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να προβάλλει κάτι αντίστοιχο. Ως προς το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, τον Οκτώβριο και Νοέμβριο θα συναντηθούμε εκ νέου και θα προσδώσουμε μεγάλη σημασία, μεγαλύτερη σημασία σε αυτό το σκέλος, σε αυτό το θέμα. Το κοινοβούλιο μας ενέκρινε την σχέση οικονομικής, ε, τη συνεργασία οικονομικής και εταιρική σχέσης Πρόκειται για μια συμφωνία η οποία θα μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή. Ίσως θα πρέπει να συγκροτηθεί μια μικτή, ένα μεικτό συμβούλιο φιλίας για να παρακολουθήσει τα θέματα ενέργειας στον ε, τομέα αυτό της εταιρικής συνεργασίας ή να δημιουργηθεί μια επιτροπή ad hoc έτσι ώστε να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία έμπρακτα. Ως προς τον διάλογο μεταξύ Σιητών και Σουνιτών, όπως σας είπα, δεν υπάρχει θέμα ε, ε σύραξης ή εσωτερικής ρήξης, αλλά ένα θέμα καθαρά διαχείρισης. η εσωτερικης ρηξης αλλα ενα θεμα καθαρα διαχειρισης στις εκλογές. Ίσως έχουμε και μια κοινή εκλογική πλατφόρμα ή κοινού εκλογικούς καταλόγους. Αυτοί οι εκλογικοί κατάλογοι και συμφωνίες είναι συμφωνίες ε, στις οποίες, οι οποίες θα, θα επέλθουν πριν από τις εκλογές, δηλαδή θα συμφωνηθούν όλα αυτά πριν από τις εκλογές για κοινού εκλογικούς ε, καταλόγους. όπου θα συμμετέχουν όλοι, όλες οι πλατφόρμες και όχι μόνο οι θρησκευτικές, ε, τα, θρησκευτικά και which we have got, you know, are very important to us. Uh, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ σημαντική η επίσκεψή σας. Ευχαριστούμε για την παρουσία και όλη την προσωπία σας. Από το Ιράκ θα ήθελα να πω ότι σας ε, διαβεβαιώνω πως θα μεταφερθούν ε, τα όσα μας είπατε και στον κύριο Μπρόκ, τον Προεδρό μας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζουμε καλωσορίζοντας τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, κύριο Αντιράμα, ο οποίος ε, ήρθε ενώπιον μας και θα παραμείνει μαζί μας 45-50 ε, λεπτά γιατί στις 6 ώρα ακριβώς έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Άρα στις 6 παρατέταρτο θα πρέπει να αποχωρήσει και θα πρέπει να έχει τελειώσει η συζήτησή μας προφανώ μέχρι τότε. Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την νίκη σας στις εκλογές. You know that uh, we appreciate... Επίσης, ε, μας ικανοποιεί και η ομαλή μετάβαση της εξουσίας και παράδοση της εξουσίας όπως όλες οι χώρες στην περιοχή συμπεριλαμβανομένες και της δικής μου της Ρουμανίας γνωρίζουμε ότι και στη χώρα σας υπάρχουν σκαμπανεβάσματα σε αυτό το δύσκολο δρόμο προς την εδραίωση της δημοκρατίας και της οικονομίας της αγοράς της χώρες μας. Χαιρόμαστε και εκτιμούμε πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθησαν οι εκλογές. Uh, uh, Νομίζω ότι ε, πιστεύουμε όλοι ότι θα συνεχιστεί το πνεύμα διαλόγου καθώς επίσης και η πολιτική συνεργασία. Τέλος θα ήθελα να επαναλάβουμε ε, την υποστήριξή μας για να δοθεί στην Αλβανία το συντομότερο το καθεστώς υποψήφιας χώρας και ελπίζουμε το Δεκέμβριο το Συμβούλιο να λάβει θετική απόφαση προς την κατεύθυνση αυτή. Και τώρα θα ήθελα να δώσουμε το λόγο στο Πρωθυπουργό της Αλβανίας, παρακαλώ. Αν θέλετε, ε, για ένα δεκάλεπτο, δεκαπέντε λεπτά, για να θέσετε το πλαίσιο για επόμενες ερωτήσεις των συναδέλφων, στις οποίες θα κληθείτε να απαντήσετε. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εκτιμώ το γεγονός ότι έχετε έρθει όλοι σας να ακούσετε αυτά που θα είχα να σας πω ενδεχομένω. Και το πρώτο που θα είχα να σας πω είναι ότι εκτιμούμε τη συνεχή υποστήριξη του κοινοβουλίου σας για πρόοδο της ε, αίτησης υποψηφιότητας έναξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Του λεχθέντος, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τις προηγούμενες κυβερνήσεις και τον προκάτοχό μου για τις προσπάθειές τους και τα όσα έχουν επιτύχει έτσι ώστε να φέρουν την Αλβανία πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως απομένουν ακόμα πολλά να γίνουν. Είμαι πεπισμένος ότι έχει ξεκινήσει μια νέα εποχή τώρα στην αλβανική πολιτική Στόχος μας όσο και φιλοδοξία της κυβέρνησης είναι να τερματιστεί η πολιτική παράδοση του παρελθόντος. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εγγυηθούμε συνεργητική πολιτική, διακομματική και να ανοίξουμε όσο γίνεται Ε, τις διαδικασίες ε, προς την ε, αντιπολίτευση για να προωθήσουμε την υπόθεση της υποψηφιότητας της Αλβανίας. Εχθές μόλις ψήφισε η Βουλή και με ιδιαίτερη χαρά θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το πνεύμα της συζήτησης αυτής. Από το εξής και μόνο γεγονός Υπάρχει ένα νέο πνεύμα τώρα στην Προεδρία της Βουλής και στον τρόπο διεξαγωγής των συζητήσεων. Έχει όλο το χρόνο ε, ε, στη διάθεση της αντιπολίτευσης, το περισσότερο από όσο ποτέ στην ιστορία ε, της Βουλής της Αλβανίας για να σχολιάσει το πρόγραμμα και τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης. Βεβαίως, είναι πολλές οι ανάγκες αυτή τη στιγμή της Αλβανίας, αλλά βασικές μας προτεραιότητες είναι και παραμένουν η υποβολή και η έγκριση των μεταρρυθμίσεων που χρειάζονται για το κράτος δικαίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Η ευρωπαϊκή μας πορεία και η ατζέντα μας είναι ο καταλήτης για τις αλλαγές που χρειάζεται η χώρα, θεωρούμε, αλλά και το μέσο εκείνο που θα μας επιτρέψει να ολοκληρωθεί αυτό που ονομάσαμε η Αλβανική Αναγέννηση. την οποία υποστήριξαν ένα εκατομμύριο ψηφοφόροι υπερψηφίζοντας τη Συμμαχία για μια Ευρωπαϊκή Αλβανία. Ταυτόχρονα Είμαι βαθύτατα πεπισμένος ότι αντιμετωπίζουμε προκλήσεις από τις πολύ θετικέ εξελίξεις στα Βαλκάνια, καθώς επίσης από τις σημαντικότατες εξελίξεις στη Συμφωνία Κωσυφοπεδίου Σερβίας. Είναι μια συμφωνία αυτή που ανοίγει μεγάλες προοπτικές, ένα ευρύ ερίζοντα ευκαιριών για όλους μας και κάτι που μας φέρνει αντιμέτωπους και με νέες προκλήσεις. Τερματίζονται εδώ λοιπόν όλες οι παλιές σειράξεις στην πρώην Ιουκοσλαβία και διανοίγονται νέες ευκαιρίες και δυνατότητες. Και η ειρήνη αποτελεί ένα μέσο για οικονομική και κοινωνική συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών μας και των λαών μας. Από την άλλη, με μεγάλο θαυμασμό παρατηρούμε όχι μόνο το ρόλο της ηγεσία του Κωσόβου, που σε αυτή τη διαδικασία συνεργασίας και ειρήνης, αλλά και την πρόοδο που γίνεται στο Κόσοβο προς την Ευρώπη, τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, την απελευθέρωση θεωρήσεων διαβατηρίων, πράγματα ε, εκ των Ουκάνευ ε, για αυτό το νεοσύστατο κράτος στην περιοχή. Είναι λοιπόν μια νέα ευκαιρία αυτή και πιστεύουμε ότι με τη βοήθειά σας, ιδιαίτερα τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και ε, πολλών φίλων και εταίρων της Αλβανίας και με τη βοήθεια της περιφέρειας ε, μας στην Ευρώπη θα μπορέσουμε να κερδίσουμε πάρα πολύ από το χρόνο που χάθηκε στο παρελθόν. Ως χώρα και κράτος η Αλβανία έχει μια εξωτερική πολιτική από τις πιο σταθερές, ανεπηρέαστη από εναλλαγές στην εξουσία και στην κυβέρνηση στη χώρα. Ταυτόχρονα όμως, τελευταία έχει διαταραχθεί κάπως από κάποιους εθνικιστικούς πυρετούς που θα πρέπει να παραμείνει μια δυσάρεστη περίοδος του παρελθόντος. Αυτό που μας ενδιαφέρει ε, στη νέα μας πολιτική είναι ε, να μην έχουμε καθόλου προβλήματα με τους γειτονές μας. Δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι με την πάροδο των ετών έχει επιτελέσει κάποια πρόοδο η Αλβανία. Επίσης όμως δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η φιλοδοξία της Αλβανίας είναι πολύ μεγαλύτερη Mates. από την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Και η φιλοδοξία αυτή θα μας καθοδηγήσει και προς το μέλλον εάν αποκομίσουμε όλα τα θετικά διδάγματα από τα θετικά αλλά και από τα αρνητικά του παρελθόντος. Είμαι ακράδαντα πεπισμένος ότι οι Αλβανοί μας ψήφισαν και μάλιστα με τρόπο σαρωτικό. Αυτό δεν ήταν απλώς το αποτέλεσμα της ανάγκης για αλλαγή ενός Πρωθυπουργού και να αντικατασταθεί από έναν άλλον ή ορισμένη υπουργοί από κάποιους άλλους ή μια παράταξη από άλλη παράταξη. Η ουσιαστική ανάγκη ήταν ανάγκη να αλλάξει η χώρα. Και αυτό το αποτέλεσμα μας κάνει να αισθανόμαστε όλοι μέτριοπαθείς και να ε, έχουμε επίγνωση απόλυτη του γεγονότος ότι έχουμε έρθει σε αυτή τη θέση και σε αυτό το αξίωμα όχι για αυτό που είμαστε, αλλά για αυτό που έχει ανάγκη ο κόσμος και αυτό που θεωρεί ο κόσμος ότι θα πρέπει να είμαστε εμείς υπέρ του λαού. Είναι τεράστια ευθύνη αυτή και είμαστε διατεθειμένοι να εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή και να επιτελέσουμε αυτό το έργο που περιμένει από εμάς και που μας έχει ζητήσει ο λαός της Αλβανίας στις 23 Ιουνίου. Επίσης πιστεύω από την εμπειρία μου από μια χώρα που πέρασε πολύ ε, δύσκολες περιόδους, δραματικές και τραγικές στο παρελθόν, κατά την ε, εποχή της, Σοβιε... της ε, κομμουνιστικής αυτοκρατορίας, όπου η Αλβανία είχε την πιο ομή δικτατορία και μια ταραγμένη μεταβατική περίοδο. Και τώρα αυτή η σαρωτική νίκη σημαίνει πολύ βαθιές αλλαγές και μεγάλη ανάγκη για την καθημερινή δημοκρατία. Το 1992 οι Αλβανοί ψήφισαν και πάλι σαρωτικά υπέρ μιας μεγάλης αλλαγής. Στις 23 Ιουνίου για δεύτερη φορά ψήφισαν τόσο μαζικά ε, για την ειρηνική εναλλαγή στην εξουσία, αλλά έστειλαν και ένα σαφέστατο μήνυμα. Αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι τα μεγάλα λόγια, η δημοκρατία με την υψηλή έννοια, αλλά η καθημερινότητα ε, στη ζωή των πολιτών. Αυτό χρειάζεται, εκδημοκρατισμός της καθημερινής ζωής των πολιτών. Ε, απαραίτητος. Και έχουμε έρθει τώρα εδώ για να σας ε, διαβεβαιώσουμε ότι όλα όσα κάνετε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάνει πολλά για την Αλβανία, δεν θα απομονμάται καθόλου αλλά θα αποτελέσουν μια πηγή έμπνευσης και ταυτόχρονα θα είναι για μας πάντα ένας λόγος παραπάνω, το συντομότερο να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας και να εκπληρώσουμε τα όσα ακόμα υπολείπονται έτσι ώστε η Αλβανία να καταστεί μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας και πλήρες μέλος με πλήρη δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ. Πολύ θερμητικά τόσο μας είπατε. Και η παρουσία σας εδώ αποτελεί εγγύηση ότι θα υλοποιηθούν. Έχω μια σειρά από εγγεγραμμένους στον κατάλογο. Παρακαλώ τους συναδέλφους να περιορίσουν τις ε, παρεμβάσεις του στα δύο λεπτά, ώστε να έχει την ευκαιρία και ο προσκεκλημένος μας να δώσει τις απαντήσεις στις ερωτήσεις. Και πρώτος θα είναι ο κύριος Κούκαν, πρόεδρος της αντιπροσωπείας. Και τον καλό να λάβει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είστε πολύ αυστηρός δύο λεπτά και θα πρέπει να δώσω και την ενημέρωση για τις εκλογές και να χαιρετήσω τον Πρωθυπουργό και να απευθύνω το μήνυμα εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ να είστε, να είστε αν ξεπεράσω κατά πέντε δευτερόλεπτα το χρόνο μου. Δυόμιση λεπτά λέει ο Πρόεδρος. Καταρχάς ευχαριστώ πολύ ε, και καλωσορίζω θερμά τον Πρωθυπουργό. Ε, τον συγχαίρω για την επιτυχία του, επιτυχία του πολιτικού του κόμματος στις εκλογές και νομίζω ότι είναι και δίκαιο και Αρμόζων εν προκειμένου να αναφέρουμε και να υπογραμμίσουμε τη δουλειά της κυβέρνησης αυτής στο στόχο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η πολιτική κατάσταση στην Αλβανία ασφαλώς ε, επικεντρώθηκε στην πρόοδο προς τη ευρωπαϊκά όργανα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση το τελευταίο διάστημα και πιστεύω ότι και η νέα κυβέρνηση που σχηματίζεται τώρα θα δώσει έμφαση σε, αυτή την, ε, σε αυτό το θεματολόγιο. Στις 23 Ιουνίου λοιπόν έγιναν εκλογές πάρα πολύ σημαντικές για την Αλβανία, εκλογές οι οποίες αποτέλεσαν δοκιμασία για το κατά πόσον και κριτήριο για τα πόσον μπορούν να εισαχθούν δημοκρατικά ε, κριτήρια και ε, για το κατά πόσο είναι αρκετά όρημα τα πολιτικά κόμματα ώστε να αποδείξουν ε, την ετοιμότητά τους ε, να ξεκινήσουν τον δρόμο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Τολμώ να πω ότι πέρασε αυτή τη δοκιμασία επιτυχώς η Αλβανία και πιστεύω ότι και στο μέλλον θα δούμε περισσότερες απτές αποδείξεις για το γεγονός αυτό. Ε, έχουμε τέσσερις συναδέλφους εδώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έλαβαν μέρος στην αντιπροσωπεία ad hoc παρατηρητών ε, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γίναμε δεκτοί με μεγάλη ευγένεια και θέρμη ε, διαπιστώσαμε ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ήταν πρώτη στην, ε, στις προτεραιότητες και στην θεματολογία αυτής της προεκλογικής εκστρατείας. Πολύ μεγάλη σημασία αποδίδεται λοιπόν στην, ευρωπαϊκή, ε, στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είδαμε ότι έγινε η εκλογική αναμέτρηση με τις αντιπαραθέσεις Φυσικά δεν μπορούμε να πούμε ότι τα πάντα κύλησαν απρόσκοπτα, θα ήταν ψέμα αυτό. Αλλά πάντως εν γέννη κρίνονται καλές οι εκλογές και το πιο σημαντικό η μετάβαση ε, στην εξουσία έγινε κατά τρόπο πολιτισμένο ο πολιτικός ε, που ιτήθηκε απεδέχθη την ήττα του, καλωσόρισε τον νέο ναι, πρωθυπουργό με τρόπο αρμόζοντα, με μια καλή και σημνή αναφορά στις πολιτικές εξελίξεις και το πολιτικό γίγνεσθε στη χώρα. Κάτι το οποίο θέλουμε να βλέπουμε να συμβαίνει και στο μέλλον. Χωρίς πραγματικό πολιτικό διάλογο των πολιτικών δυνάμεων, όλων των πολιτικών δυνάμεων στην Αλβανία, θα είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσει η χώρα. Οι εξελίξεις μέχρι τώρα δείχνουν ότι αυτό είναι δυνατόν, ότι η νέα κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να το πράξει. Στην, ε, στο πρόγραμμα της, ε, του νέου κοινοβουλίου μία από τις πρώτες θέσεις κατέχει η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω ότι θα μπορέσετε να υλοποιήσετε αυτούς τους στόχους. Βλέπω ότι δεν έχω πολύ χρόνο. Ε, το μήνυμά μου κύριε Πρωθυπουργέ είναι Χαίρομαι που σας βλέπουμε εδώ. Είστε πολύ νέος ε, στα καθήκοντά σας. Μόλις μερικές ημέρες τώρα έχετε αναλάβει καθήκοντα. Αλλά πιστεύω ότι θα μπορέσετε να εξηγήσετε και σε μας εδώ και σε όλα τα θεσμικά όργανα. Ε, δεν χρειάζεται να επαναλάβω αυτά τα οποία είπατε και εσείς, ε, ήσασταν πολύ πιστικός, αλλά πάντως σας ευχαριστώ γιατί αναφέρατε ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πολύ μεγάλη θέρμη σας υποστήριξε σε αυτή την ε, προσπάθεια για την πρόοδο στη χώρα σας. Θα συνεχίσουμε, σας διαβεβαιώνω, θα συνεχίσουμε και εμείς στο μέλλον να σας υποστηρίζουμε. Παρακαλώ λοιπόν να ε, ζητάτε όποτε ε, υπάρχει ανάγκη και όποτε είναι δυνατόν τη δική μας βοήθεια θα σας την προσφέρουμε ευχαρίστω. Ευχαριστώ κύριο Σαλαφράγκα, έχει το λόγο. Eh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα μιλήσω ισπανικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Κύριε Πρωθυπουργέ, εξ ονόματος του ΕΛΚ θα ήθελα να σας ε, καλωσορίσω, να σας συγχαρώ για τα αποτελέσματα των εκλογών και να σας ευχαριστήσω για τον επικοδομητικό και συμφιλιωτικό τόνο που χρησιμοποιήσατε σε σχέση με την αντιπολίτευση και βεβαίως ε, εδώ μιλώ για την στάση που κρατήσατε στο Εθνικό σας Κοινοβούλιο με βάση την νίκη σας και πώς αντιμετωπίζετε το μέλλον. Ε, μιλάμε για την ευρωπαϊκή ε, προοπτική της χώρας σας μέσα στα πλαίσια του νέου καθεστώτος θεωρήσεων και της προοπτικής προσχώρησης. Όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι με βάση τη μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη υπάρχουν οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο, για μια προενταξιακή διαδικασία, αλλά θα ήθελα να διατυπώσω μια ερώτηση τώρα που από αντιπολίτευση είστε συμπολίτευση, πώς θα αντιμετωπίσετε την χώρα σας για την μελλοντική ένταξη της χώρας σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορέσετε να συνεργαστείτε με την αντιπολίτευση για αυτό το μεγάλο σχέδιο. Θα σεβαστείτε τα δικαιώματα των ε, μειονοτήτων ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φλέκενστάιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, και εμείς σας καλωσορίζουμε θερμά. Σας συγχαίρουμε θερμά για τις ε, εκλογές σας, για την επιτυχία σας στις εκλογές. Και με μεγάλη χαρά σας βλέπουμε εδώ. Αναφέρατε κι εσείς μια σειρά από σημαντικά καθήκοντα, την επικράτηση του κράτους δικαίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς. Θα ήθελα κι εγώ να πιέσω λίγο ακόμα από πλευρά μου και να ρωτήσω το εξή. Εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε ώστε να ανθαρρύνουμε και εσάς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή την ε, προσπάθεια και να σας υποστηρίξουμε στις προσπάθειες σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν είχατε κάτι να προτείνετε, τι θα ήταν. Κύριε uh, Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρία Υπουργέ, εξ ονόματος της ε, ομάδας μου θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω που προσήλθατε για να συζητήσουμε και να μας μιλήσετε για τις απόψεις σας ως προς την παρούσα κατάσταση της χώρας και τις μελλοντικές εξελίξεις. Όπως είπαν και άλλοι προλαλήσαντες, η πολιτική αυτή μετάβαση, οι πολιτικές μεταβάσεις, ιδιαίτερα σε χώρες όπου ο πληθυσμός έζησε κάτω από πολιταρχικό ή δικτατορικό καθεστώς αντιμετωπίσουν μεγάλες δυσκολίες. Και βεβαίως ε, η, το να μοιράζεται κανείς την εξουσία είναι επίσης πολύ δύσκολο. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη σαρωτική αυτή νίκη και μας αναφέρετε ότι στην ε, συζήτηση στο Κοινοβούλιο μετά από την ανάληψη των καθηκόντων σας και την ορκομοσία ε, μιλήσατε για τις σχέσεις με την αντιπολίτευση. Ε, υπάρχει βεβαίως ε, και η ποροπτική μιας νέας εποχής που διανοίγεται. Γι' αυτό υπήρχε και αυτή η εφορία. Πώς βλέπετε τις σχέσεις της κυβέρνησής σας με άλλες πολιτικές δυνάμεις στη χώρα σας και με την κοινωνία των πολιτών. Έχει κλείσει ο κατάλογος των ομιλητών. Ο Τσάλς Τάνοκ έχει το λόγο. Και πάλι συγχαρητήρια εξ ονόματος της ομάδας μου των Ευρωπαίων Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών και, μετά, ε, και ιδιαίτερα μετά από τους κλειδονισμούς που γνωρίσατε τελευταία ε, ε, διετία έγινε μια ομαλή μετάβαση της εξουσίας. Ο Σάλι Μπερίσα έκανε δηλώσεις ιδιαίτερα στα Σκόπια σε σχέση με την Μεγάλη Αλβανία. Εγώ είμαι και φίλος της Μακεδονίας όπως γνωρίζετε και θα ήθελα να ξέρω ότι δεν θα αμφισβητήσετε τα σύνορα αυτής της χώρας. Ως προς τις νομιλίες βελιγραδιου Βελιγραδίου-Πρίστινα, οι συζητήσεις είναι πολύ θετικές. Πώς βλέπετε να διαγράφεται η κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια, ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών. Και ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας ως προς την οικονομική ανάπτυξη και τα επενδυτικά σας σχέδια. Τέλος, η Αλβανία ε, ε, είναι πλήρες μέλος της διάσκεψης Ισλαμικής Συνεργασίας και όπως ξέρετε πολλές φορές γίνεται διαφορετική, ακολουθείται διαφορετική θέση σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πώς βλέπετε αυτή σας τη στάση σε σχέση με την ε, μελλοντική προενταξιακή σας πορεία. Πρόεδρος, ε, θα πρέπει οι επόμενοι ομιλητές να μιλήσουν για 1,5 λεπτό πλέον για να μας απαντήσει και ο Πρωθυπουργό. Ο κύριος Πέτερλε έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε θα δείτε πόσο σύντομος ε, μπορεί να είναι ένας βουλευτής. Να σας συγχαρώ κύριε Πρωθυπουργέ, σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Κατανοώ ότι από πολιτικής ε, πλευράς θέλετε να ακολουθήσετε μια ενωτική πορεία με την αντιπολίτευση και επιζητάτε αυτή τη συνεργασία με την αντιπολίτευση. Πώς ε, θεωρείτε ότι μπορεί να προωθεί αυτή η συνεργασία κατά το μέγιστο δυνατόν. Ο κύριος Μποστινάρου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν χρειάζεται να τονίσω πόσο ευτυχής είμαι, διότι βλέπω τον φίλο μου, τον Έντι Ράμα Πρωθυπουργό, καθώς και την Υπουργό Εξωτερικών. Πέρα όμως από τα προσωπικά μου συναισθήματα, θα ήθελα να σας πω ότι ως Ρουμάνος και ως φίλος της Αλβανίας, και επειδή είμαι προευρωπαϊστής θεωρώ ότι η Αλβανία βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι και μπορεί να αλλάξει το μέλλον της. Και είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνησή σας θα ε, κάνει, θα, θα προωθήσει αυτή τη διαφορά και θα σας δοθεί το πράσινο φως για διαπραγματεύσεις για την ενταξιακή σας πορεία, στην οποία θα φτάσετε. Θα ήθελα να σας πω ότι η αντιπροσωπεία των σχέσεων με την Αλβανία θα είναι βασικό σας εταίρος για να σας βοηθήσουμε στην προσπάθειά σας και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι ο Πρωθυπουργό μου, ο Βίκτορ Πόντα, θεωρεί ότι η Ρουμανική κυβέρνηση θα είναι ένας ε, πολύ κοντινός εταίρος και φίλος όταν ε, το επιθυμείτε. Ελπίζω να επισκεφτείτε τη χώρα μου στο εγγύς ε, μέλλον και να είναι ένα νέο μια νέα ιστορική στιγμή στις διμερείς μας σχέσεις που διανύουν το εκατοστό έτος συνεργασίας. Η κυρία Πακ από το ΕΛΚ. Κύριε Πρωθυπουργέ, συγχαρητήρια. Σας εύχομαι καλή επιτυχία ε, στην εργασία σας υπέρ των Αλβανών ανδρών και γυναικών. Σήμερα εκφωνήσατε εδώ μια ομιλία που ακούστηκε πολύ συμφιλιωτική, ενίοτε και σόφρον και σοφή. Ελπίζω να διέπει αυτό και το μέλλον των εργασιών σας. Επίσης, ελπίζω οι ανοησίες των εθνικιστικών τόνων των τελευταίων ημερών να πάψουν και δεν ε, εκπορεύονται μόνο από την απερχόμενη κυβέρνηση αυτή. Ελπίζω και το είδα όταν πήγατε και στο Κόσοβο να υιοθετήσετε άλλο ύφο πλέον υπέρ της ειρήνης και προς το συμφέρον της ειρήνης στα Βαλκάνια. Θα είχα μια μεγάλη παράκληση να σας απευθύνω. Αν με τη δική σας συμπεριφορά και τη συμπεριφορά της κυβέρνησής σας ε, και παρένθεση εδώ γνωρίζω πολύ καλά την Υπουργό Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, αν φροντίσετε αυτά τα έκτροπα στο κοινοβούλιο, στον τύπο, τα ε, υποτιμητικά ε, να σταματήσουν. Ε, κάθε φορά βλέπουμε δημοσιεύματα στον τύπο για την πολιτική συμπεριφορά των διαφόρων μελών των κομμάτων. Αυτό φαίνεται και μέχρι το Υπουργικό Συμβούλιο και αυτό έχει και επιπτώσεις για την εικόνα που δίνει η Αλβανία. Αν συνεχίσετε με την εικόνα και τη συμπεριφορά που δώσατε, δείξατε σήμερα εδώ, είστε σε καλό δρόμο. Και να πω κάτι ακόμα και σε σχέση με τη δική σας συμπεριφορά και άλλων. Οι Αλβανοί είναι αρκετά όρημοι και ενήλικες να μην ε, ζητάνε ε, από όλους τους ε, διπλωμάτες επιβεβαίωση. Κάντε τη δουλειά σας. Μην ρωτάτε όλους τους διπλωμάτες ε, ωραία τα κάνουμε καλά, τα πάμε. Τι δουλειά έχουν οι διπλωμάτες, δεν είναι δάσκαλοι σας. Μέχρι τώρα κάποιοι το έκαναν και εσείς το ίδιο. Παρακαλώ αυτό να σταματήσει για να δείξετε κάποια οριμότητα ότι προχωρείτε περισσότερο προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ε, σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ κυρία Γκόμες. My Καταρχήν να σας συγχαρώ και εγώ, ε, όπως ξέρετε, ο συνάδελφος μίλησε εξ ονόματος της ε, δικής μου πολιτικής ομάδας. Ελπίζω να μπορέσετε να βασιστείτε την ε, μακρά σας ε, πείρα πριν από τις εκλογές ότι θα μπορέσετε να προωθήσετε μια δημοκρατία χωρίς αποκλεισμού στην Αλβανία. Θα ήθελα να μας μιλήσετε για τις σχέσεις με τις γείτονες χώρες και ορισμένα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει σε εθνικό επίπεδο, όπως η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Όμως η καταπολέμηση της διαφθοράς δεν είναι εθνικό φαινόμενο, είναι ένα ε, διεθνικό φαινόμενο. Πώς ε, επινοείτε, μάλλον ποια είναι η στρατηγική σας και πώς θα την αντιμετωπίσετε με βάση τον τρόπο με τον οποίο την αντιμετωπίζουν και οι γείτονες χώρες. Η κυρία Γιαννάκου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας για την εκλογική του νίκη και να του ευχηθώ καλή θητεία και να σημειώσω ότι όλοι μας εδώ λίγο πολύ έχουμε υποστηρίξει την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας με διάφορες ευκαιρίες και κατά την εκπόνηση των εκθέσεών της. Ένα από τα τμήματα, μια από τις αρχές που αφορούν στις χώρες οι οποίες πρόκειται να ενταχθούν στην Ένωση είναι η σχέση καλής γειτονίας και βέβαια πολύ περισσότερο η σχέση καλής γειτονίας με τις χώρες της Ένωσης. Ήθελα να σας ρωτήσω κύριε Πρόεδρε, το 2008 η κυβέρνηση Μπερίσα για την οποία είπατε ότι λίγο πολύ είχατε την ίδια εξωτερική πολιτική έκανε μια συμφωνία με την Ελλάδα για τον καθορισμό των χωρικών υδάτων εσείς προσωπικά προσφύγατε στο δικαστήριο για να καταρρίψετε αυτή τη συμφωνία και το καταφέρατε. Νομίζετε ότι οι σχέσεις με την Ελλάδα είναι ασήμαντες ή μπορούν να κρίνονται από τα δικαστήρια και τι σκοπεύετε να κάνετε στο μέλλον για αυτή την υπόθεση που ενδιαφέρει και τις δύο χώρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τάνια Φαϊόν. Ευχαριστώ πολύ. Συμμερίζομαι και εγώ και συμφωνώ ε, με τα ε, αισθήματα και τις σκέψεις των συναδέλφων ε, και τα συγχαρητήρια. Χαίρομαι που βλέπω τόσο πολλούς γνωστούς μέλη στην κυβέρνηση και τόσο πολλούς ευρωπαϊστές. Είναι ισχυρό το μήνυμα σας ε, ε, κύριε Πρωθυπουργέ, φτάνετε στις Βρυξέλλες λίγες μόνο ώρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης. Και αυτό δείχνει πόσο προσιλωμένοι είστε στην ευρωπαϊκή πορεία της ε, χώρας. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να σπάσει η πολιτική παράδοση του παρελθόντος, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις εμπλοκές, την έλλειψη μεταρρυθμίσεων και διαλόγου που διαπιστώναμε στο παρελθόν που δεν συνομιλούσαν καν τα πολιτικά κόμματα. Όλα αυτά χρειάζονται και ακόμα περισσότερο για να κινητοποιηθεί και η κοινωνία των πολιτών και οι μη κυβερνητικέ οργανώσει και να λειτουργούν όλοι οι δημοκρατικοί θεσμοί σωστά και να ακούτε και τι ανάγκε των πολιτών. Η Αλβανία ήταν όντω η πιο απομονωμένη χώρα και πιστεύω ότι αξίζεται περισσότερο από ποτέ μια κοινωνία ανοιχτή και δημοκρατική. Και θα ρωτούσα το εξής πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το θέμα της ανεργίας των νέων, ε, πώς θα τους κάνετε να παραμείνουν στη χώρα τους οι νέοι. Και μια ερώτηση σε σχέση με αυτό που είπε η Άννα Γκόμες, η διαφορά. Αύριο ολοκληρώνουμε ε, το, τις εργασίες της ειδική Επιτροπής μας ε, και έχουμε κάποιες ιδέες για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό στην περιοχή ε, ευρύτερα, σε όλα τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μόνο αλβανικό ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Σόπφλιν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω και εγώ. Θέλετε να επιλύσετε τα προβλήματα με τις γείτονες χώρες. Αυτή είναι μία αμφίδρομη πορεία. Δεν εξαρτάται μόνο από εσά, αλλά πώς από στρατηγικής πλευράς βλέπετε να αναπτύσσετε η Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Όλοι ξέρουμε την ιστορία. Ποιος είναι ο ρόλος της Τουρκίας ή ο ρόλος του Ισλάμ και της Μέσης Ανατολής στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, πρέπει να πάρουμε σοβαρά την ιδέα της Μεγάλης Αλβανίας. Ο κύριος Λίσεκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εντάχει, Πρωθυπουργέ, κατανοείτε ότι ό,τι μας ε, λέτε για το κοσυφοπέδιο ε, παρακολουθείτε εκ του σύνεγγυς από ορισμένε χώρες, ιδιαίτερα εκείνες που δεν αναγνωρίζουν το κοσυφοπέδιο, όπως η Σερβία. Ποια είναι η θέση σας, ποια είναι η απόψή σας σε σχέση με τις μόνιμες ε, ε, συναντήσεις ε, μεταξύ μόν και του κοσυφοπεδίου. Αν κοιτάξουμε το χάρτη βλέπουμε ότι η μεγάλη σας ευκαιρία είναι ο τουρισμός. Πώς θα υποστηρίξετε αυτό το σκέλος της οικονομίας και πώς θα ανοιχτείτε στους ξένους επενδυτές. Ο κύριος Κάτιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, να σας συγχαρώ και εγώ και σας εύχομαι κάθε επιτυχία Ελπίζω να μπορέσετε να φτάσετε σε, στις διαπραγματεύσεις, στην έναρξη διαπραγματεύσεων για την ε, προενταξιακή σας πορεία και την ε, ένταξη στη συνέχεια. Ορισμένα χρόνια πριν, κατά τις εκλογές, τις προηγούμενες εκλογές, μας είπατε ότι φοβόσαστε ήταν ότι θα υπήρχε ε, διαφθορά ή θα μπορούσε να χρηματιστούν μέλη ακόμα και του δικού σας, ε, της δικής σας λίστας αν αποκαλύπτατε τα ονόματά τους ε, εγκαίρως. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε ποια είναι η δική σας άποψη και πώς θα καταπολεμήσετε τη διαφθορά στο ίδιο σας το κόμμα καταρχήν. Ας μην ε, μιλήσουμε για την αντιπολίτευση. Ο καθένας πρέπει να αντιμετωπίζει τα του οίκου του πρώτα. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αισθάνομαι καταρχάς ιδιαίτερη τιμή για το ασύνθεσο αυτό ενδιαφέρον για μια χώρα μικρή και για έναν νέο στη θέση αυτή πρωθυπουργό, όπως είπε ο κύριος Κούγκαν. Θα ήθελα να ευχαριστώ όμως και τον κύριο Κούγκαν και τον κύριο Προστινάρο για την καταπληκτική δουλειά και την καταπληκτική υπομονή που έδειξαν σε όλους εμάς στην Αλβανία. Μπορεί να δημιουργεί ε, λόγους ανησυχίας η χώρα αυτή, αλλά ποτέ δεν είναι βαρετή. Η Doris Pack, να, τόσα χρόνια ασχολείται με την περιοχή και παραμένει νέα. Σε ευχαριστούμε πολύ Doris που δεν έχεις εγκαταλείψει τον αγώνα. Και επιτρέψτε μου, στο βαθμό που μπορώ, να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Ξεκινώ με κάτι το οποίο για μένα αποτελεί την έκφραση της φιλοδοξίας μας ε, για την ε, Αλβανία. Η κυβέρνησή μας έχει το μεγαλύτερο αριθμό γυναικών από όλες μαζί τις ε, κυβερνήσεις στην περίοδο αυτή της μετάβασης που κρατάει τόσο καιρό. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την υποστήριξη. Έχουμε γυναίκα υπουργό ε, κοινωνικής ε, ε, ένταξης και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ε, εξωτερικών. Κάτι που είναι μάλλον ασύνηθες. Θα ήθελα επίσης να πω ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό και για το πώς βλέπουμε το μέλλον μας. Το μέλλον της συνεργασίας και το μέλλον των συνόρων. Στις 23 Ιουνίου αγωνιστήκαμε και κάναμε τις εκλογές με τη Συμμαχία για την Ευρωπαϊκή Αλβανία όπως την ονομάσαμε και μας τίμησαν οι πολίτες με ένα εκατομμύριο ψήφους. Αποτέλεσμα άνευ προηγουμένου, ενώ το εθνικιστικό κίνημα δεν έλαβε ψήφους, ένα εθνικιστικό κίνημα το οποίο εμφανίστηκε στο πολιτικό σκηνικό και προκάλεσε ταραχές, έμεινε εκτός κοινοβουλίου. την πεποίθησή μου είναι πως ένας από τους λόγους από τους οποίους το Δημοκρατικό Κόμμα, όπως ονομάζεται, έλαβε τόσο κακά αποτελέσματα ήταν και διότι παρεξέκλεινε προς ορισμένες εθνικιστικές τοποθετήσεις, τοποθετήσεις απαράδεκτες και για την εποχή μας, αλλά και για τις θέσεις που θα εξέφρασε κανείς ε, εκ μέρους της Αλβανίας προς τους φίλους και γείτονες, αλλά εξίσου απαράδεκτες και για το ε, μέλλον και τις προοπτικές της χώρας. Είμαστε πεπιθυσμένοι ότι υπάρχουν σύνορα τα οποία όμως δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν εμπόδιο σε μια συνεργασία και ενότητα όχι μόνο για τους Αλβανούς τους ίδιους, αλλά και για τη σχέση των Αλβανών με τους Σέρβους, τους Μαυροβούνιους, τους Βοσνίους, αλλά και τους Κροάτες αργότερα όταν ε, φτάσουμε να συστήσουμε ευρύτερα και τους Έλληνες και τους Ιταλούς και τους Τούρκους. Εξού και η συμφωνία Αλβανίας Κοσμοπεδίου είναι ε, μεταξύ Σερβίας Κοσμοπεδίου αποτελεί την, ε, το τέλος μιας εποχής, σημειοδοτεί το τέλος μιας εποχής και μιας μεγάλης σύγκρουσης και από εδώ και προς πρέπει να δούμε τι θα την κάνουμε. Θα συνεχίσουμε να είμαστε οι ταραχοποιοί για τις Βρυξέλλες. Θα έχουμε κάθε φορά κάποιες υποδείξεις για το πώς θα κάνουμε τα μαθήματά μας ή πια θα αρχίσουμε να χαράσουμε το μέλλον μας και να θέτουμε στόχους. Και καθώς πολύ σωστά οι Βρυξέλλες μας καλούν και μας προκαλούν να ε, κάνουμε το έργο μας, θα πρέπει και εμείς να καλούμε και να προκαλούμε τις Βρυξέλλες με μεγάλα εγχειρήματα, με σχέδια, με βήματα συγκεκριμένα για την ειρήνη, με την απέτηση για μια υποστήριξη οικονομική και κοινωνική, κυρίως για τις επόμενε γενιές. Γιατί μπορούμε να μιλάμε για το σήμερα κάθε μέρα, ταυτόχρονα όμως όποιος ε, γεννήθηκε αμέσως μετά το πέρας του κομμουνιστικού κοθιστότος, τώρα πια σχεδόν ετοιμάζεται να κάνει παιδιά. Άρα λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον. Και βλέπουμε ότι χρειάζεται πολύ περισσότερος εξευρωπαϊσμός και αντίληψη ηθαγένειας, ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Αυτό δεν θα το παρεμποδίσουν σύνορα. Μόνο η φραγμή μέσα στο μυαλό του καθενός. Η φραγμή που κατά κάποιο τρόπο μας έχει αφήσει ως παρακαταθήκη ιστορία που δεν ήταν τόσο γενναιόδορη με μας. Συχνά και δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν κομμουνιστή ενδεχομένω παρόντα. Ε, συχνά οι κομμουνιστές στρέφονται κατά των ανθρώπων και όχι των επιχειρημάτων. Καταπολεμούν ανθρώπους και όχι επιχειρήματα. Αυτό που συνέβη λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια και μετά την πτώση του κομμουνισμού ήταν ακριβώς μια σύγκρουση στηριζόμενη στο ε, άλλο ως εχθρό που προσπαθούσε να καταπολεμήσει τον άλλον ως εχθρό και όχι κάποιες ιδέες, να όχι να δώσει επιχειρήματα και ιδέες. Αυτό λοιπόν θα είναι και ένα από τα πρώτα μας ε, έργα. Η συζήτηση μέσα στον κυβερνητικό μας, ε, στο κυβερνητικό μας συμβούλιο ξεκινάει όχι με κάποιο αίσθημα εφορίας, αλλά με το καθήκον και το εργαλείο που θα πρέπει να ετοιμάσουμε και με το οποίο θα πρέπει να ε, απευθυνθούμε στο Κοινοβούλιο για να το εγκρίνει και για να δείξουμε στην ε, ε, αντιπολίτευση ότι εμείς ό,τι έχουμε ζητήσει ως αντιπολίτευση θα το διεκδικήσουμε. Όπως άλλωστε και εδώ σοσιαλιστής πρόεδρο στην Επιτροπή πάντα είναι πολύ πιο επίοικη ω προ το χρόνο ομιλία από ότι είναι συντηρητικό ε, πρόεδρο. Πάντα είναι καλύτερο λοιπόν να υπάρχει σοσιαλιστή πρόεδρο, λέει ο μιλητή. Αυτά είχα να πω για τον εθνικισμό και τα σύνορα. Και θα ήθελα να πω και κάτι ακόμη. Η Αλβανία είναι μια χώρα η οποία έχει και φυλάτη έναν πολύτιμο θησαυρό της, πολιτικ... της ε, ανεξιθρησκείας και της απρόσκοπτης συμβίωσης μεταξύ Ορθοδόξων, Καθολικών, Μουσουλμάνων. Ε, είτε πρόκειται για μουσουλμάνο, είτε πρόκειται για χριστιανό, ορθόδοξο, καθολικό. Εμείς δεν βλέπουμε τον άνθρωπο με γνώμονα τη θρησκεία του, αλλά μόνο ως άνθρωπο. Αυτό σεβόμαστε και αυτό θέλουμε να διφυλάξουμε. η περιοχή μας η ευρύτερη υποφέρει ακριβώς από αυτό. Από το να χαρακτηρίζεται κάποιος ως μουσουλμάνος ή ως χριστιανός. Όταν αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τον συγκεκριμένο άνθρωπο και το Θεό του. Και με αυτόν πρέπει να το λύσει. Όχι με τους υπάλληλους ανθρώπου του. Αυτό λοιπόν είναι η δική μας θεώρηση και έτσι δεν ε, βλέπουμε ούτε κανένα εμπόδιο προς το να συμμετάσχει η Τουρκία ως στρατηγικός εταίρος μαζί με την Ιταλία και την Ελλάδα. Τουναντίον ε, θεωρούμε ότι μπορούμε να καλύψουμε και ένα κενό της πολιτικής μας, του παρελθόντος, εξωτερικής μας πολιτικής του παρελθόν, ε, προχωρώντας αυτό το βήμα. Έτσι λοιπόν, με τρεις στρατηγικούς εταίρους, μπορεί η Αλβανία να βρει τη θέση της και μέσα στην περιοχή και να εργαστεί για το καλό όλης της περιφέρειας. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος του αντίον θα έπρεπε η κυβέρνηση της ε, Αλβανίας μαζί με την κυβέρνηση του Κοσμοπεδίου να συνεργαστούν. Αν συνέβαινε το ίδιο ε, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, φανταστείτε πώς θα ήταν. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να συζητήσουν για το μέλλον, για τη συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών, για την περιφερειακή συνεργασία, για τα οικονομικά, τα κοινωνικά ε, σχέδια, την ε, παιδεία, τον πολιτισμό. Όλο αυτό το ευρύ φάσμα ευκαιριών που θα πρέπει να διεκδικήσουμε και να υλοποιήσουμε. Ας μην μείνουν λοιπόν ε, που κάμισα διανό αυτές οι εξαγγελίες, ας τις καταστήσουμε ουσιαστικές, ας τις συμπληρώσουμε με το ευρωπαϊκό όραμα για να μην αφήσουμε πεδίο κενό, πεδίο στο οποίο θα μπορούσαν να εμφανιστούν εθνικισμοί, ε, αισθήματα, ε, αισθήματα διάψευσης και ματέωσης και εντάσεις. Και θα ήθελα να σας επισημάνω το εξής. Πολλοί πιστεύουν ότι ανεξάρτητο Κόσοβο και χωριστεί ο κράτος Αλβανίας θα μπορούσε να αποτελέσει καταστροφική εξέλιξη για την περιφέρεια. Όχι, το αντίθετο θα ήταν ε, λάθος. Όπως ε, λάθος και ανοησία ήταν το να μην αναγνωρίσετε το Κόσοβο. Και αυτό πιστεύω ότι η πλήρης αναγνώριση του κοσμοπεδίου μέσα στην Ευρώπη, ως χώρα μέσα στην Ευρώπη, όχι μόνο είναι κάτι το σωστό, το ορθό και φόρος στην ιστορία των ανθρώπων, αλλά σωστό και συμφέρον και για την ε, περιφέρεια ολόκληρη και για την Ευρώπη. Προχωρώντας, θα ήθελα να πω ότι ταυτόχρονα ακράδαντα ότι η διαφορά και το οργανωμένο έγκλημα, όπως είπε και η κυρία νωρίτερα, δεν είναι κάτι το εθνικό, είναι διεθνές φαινόμενο. Όπως η διαφήμιση της Νόκια, ξέρετε, συνδέει τους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν, connecting people, θα πρέπει να αγωνιστούμε για εξυγχρονισμό, για συνεργασία, για κοινή αντιμετώπιση. Η σωστή απάντηση στη διαφθορά είναι ο εξυγχρονισμός. Ο εξυγχρονισμός των κρατικών δομών, των κρατικών υπηρεσιών, των κρατικών φορέων. Η διαφθορά επικρατεί και ανθεί εκεί όπου μπορεί να προσφέρει μια εναλλακτική, γιατί κάτι λείπει και δεν έχει μια υπηρεσία σωστή ο πολίτης. Η δε ενδυμική διαφθορά που χαρακτηρίζει και ταλανίζει την Αλβανία ακριβώς σε αυτό το φαινόμενο οφείλεται, στο ότι η διαφθορά αποτελεί εναλλακτική ε, και καλύπτει το κενό υπηρεσιών, φορέων, κρατικών δομών που απουσιάζουν, που λείπουν. Γιατί δεν υπάρχουν οι δομές και οι υπηρεσίες που χρειάζεται ο πολίτης, στο επίπεδο του πολίτη. Ο νέος Υπουργός Κοινωνικής Ο νέος υπουργός, η νέα Υπουργός Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης έχει φιλόδοξο πρόγραμμα. Θα έχει όλη μας την υποστήριξη και αυτό το εννοώ όχι μόνο μεταξύ κομμάτων αλλά και σε στενή συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης, κομμάτων και κοινωνίας ώστε ολόκληρο το έθνος ως ένα σώμα να υποστηρίξει την, το τα ευρωπαϊκά εδεώδη και την ευρωπαϊκή ολοκληρώση και ένταξη στην Ευρώπη ως διαδικασία. Και πιστεύω ότι όπως, ε, εάν, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν, μείνει στο περιθώριο, ε, αποκλειστεί από αυτές τις διαδικασίες η αντιπολίτευση και μετατραπεί η κοινωνία των πολιτών σε μια πελατειακή κοινωνία, η οποία έχει ήδη κάνει μεγάλο κακό και θα εξακολουθήσει να ζημιώνει τις προσπάθειές μας, ε, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αυτό θα σταματήσει λοιπόν, θα πάψει και θα πάψει εδώ και τώρα. Είναι σημαντικέ οι μεταρρυθμίσει που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν. Αλλά ένα πράγμα πρέπει να υπογραμμίσω για να το γνωρίσετε και εσεί και όλοι. Ότι η πλειοψηφία είναι οριακή ειδική πλειοψηφία ή ενισχυμένη πλειοψηφία, δηλαδή η πλειοψηφία που χρειάζεται για να ε, περάσουν όλες οι, όλοι οι νόμοι που συνεπάγεται η προσπάθεια για την ένταξη. Δεν θα σταματήσουμε όμως εκεί. Δεν θα αγωνιστούμε για τη μία ψήφο που μπορεί να μας λείψει. Ξέρετε ότι αυτό δεν είναι δύσκολο, το, το γνωρίζετε κι εσείς από, ιδιαίτερα από τις ε, πρώην χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, αλλά εμείς θα το ξεπεράσουμε αυτό το επίπεδο, γιατί υπάρχουν μεταρρυθμίσεις που μπορούμε από κοινού να προωθήσουμε και θα ακούσουμε, θα αφουγκραστούμε, αλλά θα διατηρήσουμε την ιδιωτική μας θέση. Δεν θα περιοριστούμε στο να ακούμε, στο να αφουγκραζόμαστε, θα καλέσουμε, θα καλέσουμε τον κάθε έναν να συμμετάσχει, Ταυτόχρονα όμω εμεί θα διατηρούμε στα χέρια μα, θα κρατάμε στα χέρια μα το πυρδάλιο και θα επιταχύνουμε ακόμη περισσότερο για να κερδίσει το χαμένο έδαφο η χώρα. Ε, Διοικητικέ μεταρρυθμίσει πρέπει να γίνουν. έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό δήμων και κοινοτήτων που συνοδεύεται από ένα τεράστιο προπολογισμό, κονδύλια που δαπανώνται για την ε, λειτουργία μιας πολύ δυσλειτουργικής τοπικής αυτοδιοίκησης, που ταυτόχρονα ε, ε, διατηρεί αυτό το σύστημα της διαφθοράς. Υπάρχουν φωνές και από την αντιπολίτευση, τις οποίες θα, ακούσουμε, προσεκτικά. Θα καλέσουμε να συμπορευτούν μαζί μας και άνθρωποι από την αντιπολίτευση όπου έχουν εκφράσει θέσεις σωστές και παρακολουθούμε πάντοτε κάθε βήμα πολύ προσεκτικά και με επαλήθευση των ε, στόχων. Θέλουμε μια μεταρρύθμιση που θα στηρίξουν και θα ε, προωθήσουν όλοι οι πολιτικοί φορείς. Έχουμε ε, διαφορετική εικόνα στα αστικά κέντρα με ε, νέους οικισμούς, ε, παράνομες αφαίρετα οικήματα, εγκαταστάσεις χωρίς αδειοδότηση που πρέπει να νομοποιηθούν, που πρέπει να βρουν λύσεις. Έχουμε αγρότες που δουλεύουν τη γη χωρίς να έχουν πράξη κτηματολογίου που να αποδεικνύει την κυριότητα στη γη αυτή. Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε για να μετατρέψουμε την Αλβανία. Όταν πολλοί είναι αυτοί ε, ή κάποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ζητούν να μετατρέψουν τη χώρα σε μοναρχία και όταν εκλογές γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια, ξέρουμε ότι είναι περιορισμένος ο χρόνος που έχουμε στη θέση μας, πρέπει να δουλέψουμε πολύ γρήγορα και ξέρω ότι προς το συμφέρον των πάντων είναι να υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι. Για να ολοκληρώσω και ελπίζοντας ότι έχω δώσει απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, θα ήθελα να δώσω την απάντηση στην Ελληνίδα, συνάδελφο και φίλοι... για να πω για άλλη μια φορά πως η εξωτερική μας πολιτική είναι πολιτική μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες και υπάρχουν στη διάθεσή μας όλα τα μέσα για να επιλύσουμε προβλήματα που μας έχει αφήσει το ιστορικό παρελθόν. Υπάρχουν σαφέστατες δηλώσεις από πλευράς μας όλους αυτούς τους μήνες κατά των εθνικισμών, κατά του εθνικισμού και μάλιστα και σε χρονική στιγμή όπου κινδυνεύαμε να χάσουμε την υποστήριξη των ψηφοφόρων ή κάποιες ψήφους. Ε, ξεκάθαρα δηλώσαμε ότι είμαστε κατά του εθνικισμού και τώρα ως κυβέρνηση δηλώνουμε ότι είμαστε μια κυβέρνηση προσανατολισμένη απολύτως και πλήρως στην ευρωπαϊκή πορεία μας. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Είμαι όμως απολύτως πεπισμένος ότι θα έχουμε τη δική σας υποστήριξη. Και για να κλείσω με την ερώτηση στην οποία, την οποία μου κάνατε, τι άλλο θα μπορούσατε να κάνετε για να σας υποστηρίξετε, το μόνο που μπορώ να πω είναι συνεχίστε όπως κάνατε μέχρι τώρα, επηρέασε πολύ θετικά, επέδρασε πολύ θετικά η δική σας τοποθέτηση και οι ε, κινήσεις του Κοινοβουλίου, το οποίο επηρεάζει πολύ από ό,τι φαίνεται την κοινή γνώμη της Αλβανίας. Σας διαβεβαιώ ότι η φωνή σας θα ακουστεί ακόμη πιο δυνατά και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Minister, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρωθυπουργέ. Ε, όπως ε, είπαμε γνωρίζετε ότι μπορείτε να προσβλέπετε στην υποστήριξή μας και τώρα έχετε άλλη ανημενή υποχρέωση. Αν μου επιτρέπετε, ο Υπουργός Εξωτερικών ε, μου λέγει ότι δεν απάντησα στην ερώτηση για τη Μακεδονία. Ε, αν είστε φίλος της Μακεδονίας, είστε και φίλος της Αλβανίας και η εδαφική ακαιρεότητα της Μακεδονίας είναι εξίσου σημαντική για μας με την ε, εδαφική ακαιρεότητα της Αλβανίας. Ευχαριστώ.